κόμμα προς το οποίο να απευθυνόμαστε και που συζητούμε. Και να θυμάστε ότι αυτό που διακυβεύεται εδώ είναι η πιο στενή επαφή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενώσης και της Ουκρανίας. Ευχαριστώ κύριε Μιχάλσκι. Ο κύριος Κάμπελ Μπάνγκημαν έχει το λόγο. Για ένα λεπτό. Κύριε